Um, Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Ξεκινάμε λίγο πιο αργά από ό,τι συνήθως, ε, διότι δεν ε, θα συζητήσουμε το πρώτο σημείο. Περνώ σε ανακοινώσει του Προέδρου και μετά θα μιλήσουμε για την επιχείρηση Σοφία και μετά θα περάσουμε στις ψηφοφορίες. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τι ανακοινώσει του Προέδρου, καταρχά, ε, έγκριση τη ημερησία διάταξη, έχουμε τρει αλλαγέ. Το σημείο 4, που ήταν η ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι τρέχουσε διαπραγματεύσει με Αίγυπτο, Ισραήλ, Αλγερία, Ιορδανία, Λίβανο, Μαρόκο, την Ισία και Τουρκία σε σχέση με διεθνεί συμφωνίε για την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με την Europol, αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίασή μα στι 11 Απριλίου. Το σημείο 7, που ήταν η έγκριση του σχεδίου γνωμοδότηση για τη σύναψη συμφωνίας αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση με την ΕΚΑΧ αναβάλλεται και αυτό για τις 11 Απριλίου. Το σημείο 9 επίσης έγκριση του σχεδίου έκθεσης για κοινά πρότυπα και διαδικασίες στα κράτη-μέλη για τις επιστροφές, αναδιατύπωση, αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση και αυτό στις 11 Απριλίου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Εγκρίνεται όπω τροποποιήθηκε η μερίσια διάταξη. Σε ό,τι αφορά το γλωσσικό καθεστώ, έχουμε όλε τι γλώσσε πλην δανέζικων, κροατικών, μαλτέζικων και ιρλανδικών. Κατά εξουσιοδότηση και εφαρμοστικέ πράξει, 27 Μαρτίου, 2 αντιρρήσει και καταθέσει επιτροπή μα προ την ε, κατά εξουσιοδότηση πράξη Κομισιού που τροποποιεί τον κανονισμό. Κάτι θόρυβο υπάρχει, τέλο πάντων για τροποποίηση λοιπόν του κανονισμού που θεσπεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ιστορική Ασφάλεια μέσο χρηματοδοτική υποστήριξη για τα εξωτερικά σύνορα και τι θεωρήσει και σε ό,τι αφορά την κατεξοδότηση πράξη που τροποποιεί τον κανονισμό για το Ταμείο Μετανάστευση Ασύλου, κρίθηκαν το λαμέλι σε σαφή ε, πλειοψηφία στην ψηφοφορία. Δεν μπορούν λοιπόν οι δύο αυτέ ε, αποφάσεις της Κομισιόν να εγκριθούν. Θα έχουμε στις 4.30 ψηφοφορίες, οπότε σας παρακαλώ να έχετε έτοιμες και τις ε, κάρτες της ψηφοφορίας. Τέλος, πριν περάσουμε στο πρώτο σημείο της μασιάς διάταξης, Έχουμε την έγκριση των πρακτικών 6 Σεπτεμβρίου 18, 26, 27 Μαρτίου 18, 18 Οκτωβρίου 18, 29 Ιανουαρίου 19, 6 Σεπτεμβρίου 18, 26 Απριλίου 18, 27 Φεβρουαρίου 18, 20 Φεβρουαρίου 18. Εγκρίνονται αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Εντάξει, ωραία. Αγαπητοί συνάδελφοι, σημείο 9. ό,τι αφορά τη νέα εντολή για την επιχείρηση Σοφία. Είναι ένα θέμα που το έχουμε ήδη συζητήσει. Έχουμε όμως και τον Πέδρο Σεράνο εδώ από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ε, Δράσης αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή. Ζητήσαμε και από τη Ρουμανική Προεδρία εκπροσώπους, δυστυχώ όμω δεν μπόρεσαν να στείλουν κάποιον, κάτι το οποίο μα απογοητεύει. Η κατάσταση της Λιβύης είναι προτεραιότητα, ίσως ε, καλό θα τον είχαμε ακούσει ε, και από αυτούς, αλλά θα ακούσουμε από τον κύριο Σεράνου. 29 Μαρτίου αποφάσισε το Συμβούλιο να παρατείνει την επιχείρηση Σοφία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος βασική εντολή αυτή τη επιχείρηση όπω ξέρετε, είναι να συνεισφέρει στο έργο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να διαταράξει εντό αγωγικών το επιχειρηματικό μοντέλο τη διακίνηση μεταναστών και γενικώ εμπορία ανθρώπων στην Νότια Κεντρική Μεσόγειο. Οι συνάδελφοι που είναι παρόντε γνωρίζουν για την επιχείρηση Δεν θα πω λοιπόν κάτι περισσότερο για να αφιερώσουμε όλο το χρόνο που έχουμε σε, μια, σε βάθος συζήτηση με τον Πέδρο Σεράνο. Θα Παρακαλέσω λοιπόν τον κύριο Σεράνο να μας πει πόσο ο ίδιος εκτιμά την κατάσταση σε σχέση με την επιχείρηση Σοφία και θα ήθελα να μας πείτε και ορισμένα λόγια για τη γενική κατάσταση στη Λιβύη και πώς αυτή επηρεάζει τις επιχειρήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και καλησπέρα σε όλα τα μέλη της Επιτροπής σας και τους συναδέλφους βρίσκονται στην αίθουσα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ. Είναι μια σημαντική στιγμή, πολύ επίκαιρη για το θέμα αυτό. Όπω είπατε και εσεί κύριε Πρόεδρε, κατάσταση αυτή τη στιγμή στη Λιβύη και κυρίω γύρω από την Τρίπολη είναι πολύπλοκη. Οι επιχειρήσεις εκτελήσονται την ώρα που μιλάμε από τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, τον κύριο Χάφταρ. Το στρατάρχη Χάφταρ που την προηγούμενη εβδομάδα διακήρυξε την πρόθεσή του να καταλάβει την Τρίπολη. Η πατεκπρόσωπος ε, και αντιπρόεδρος Κομισιόν κ. Μογκερίνη έχει δραστηριοποιηθεί εκ τότε μετά τις δηλώσεις του Χάφταρ και συντονίζει τις δράσεις ε, μαζί με τον Γενική Γραμματέα ε, του ΕΚΕ. Συναντήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και με τους προσεξωτερικών της ομάδας των 7, G7 και κατά πιθανότητα θα συζητηθεί και στο Λουξεμβούργο στη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων πώς έχει κατάσταση. Ε, είναι πολύ ρευστά τα πράγματα και δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Έχουμε μια σαφή εικόνα της έκβασης, της κατάστασης. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύουμε και οι πρόσωποι και η ΕΔ λέμε ότι δεν μπορεί με τη χρήση βίας να βρεθεί λύση. Είναι σημαντικό λοιπόν να οι πλευρές να επανέλθουν ε, στην ε, διαπραγμάτευση υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και του ειδικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Εθνών κ. Σαλαμίου που όπως ξέρετε είχε ξεκινήσει μια διαδικασία και στις 14 Απριλίου θα ήταν η επόμενη φάση άρα προχωρούσαμε προς την εξέβρεση μιας λύσης στην τρέχουσα κατάσταση της αστάθειας στην Λιβύη. Και μια εκλογική διαδικασία που θα έδινε μια σταθερή πολιτική λύση και με συνταγματική μεταρρύθμιση. Όμως ε, οι ενέργειες ε, του στρατάρχη Χαφτάρ έχουν ε, διαταράξει αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό θα συνεχίσουν ε, να διαταράσουν και πόσο θα συνεχίσει να προελάβουν. Είχαμε αρχές της ημέρα ε, μάχες και στα προάστια ε, ένοπλες και στο αεροδρόμιο, στο Ματίγκο, στο Ιθές αεροδρόμιο που φαίνεται ότι και αυτό θα έχει πρόβλημα τελευταίες πληροφορίες. Υπάρχει έκκληση για αποκλιμάκωση ε, της ε, χρήσης βίας και θα συνεχιστούν αυτές οι εκκλήσεις από τη διεθνή κοινότητα που είναι ενωμένη και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που συνήλθε σε μια έκτακτη συνεδρίαση στο Σάββατο Κυριακό και απίφθαν και αυτό εκκλήσεις ε, σχετικά. Αυτή είναι η κατάσταση. Λύση δια της βίας δεν μπορεί να βρεθεί. Αυτό είναι σαφές. Η κατάσταση στη Λιβύη όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ ξεκάθαρα εμείς στηρίζουμε την ε, κυβέρνηση Εθνικής ε, Ενότητας ε, και αυτή η κατάσταση με τη μεμονωμένη δράση του Χαφτάρ και το Λιβικό στρατό επιπεριπλέκει τα πράγματα. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες, διότι εκτελήσεται συνεχώς η κατάσταση. Ελπίζουμε εμείς να προχωρήσει σε μια κατεύθυνση που θα δώσει δυνατότητα στη διεθνή κοινότητα να συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη αυτή τη διαδικασία που δρομολόγησε ο δικό εκπρόσωπο, αλλά και έτσι να επανέλθουν οι πλευρέ σα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, φεύγοντα από ε, το θέατρο επιχειρήσεων, ιδίω γύρω από την ε, Τρίπολη που είναι και πολυπληθή ε, ε, μια πόλη με πάρα πολλούς κατοίκους και θα έχουμε σημαντικές απώλειες αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Σε ό,τι αφορά την επιχείρηση Σοφία, η σημερινή κατάσταση με τη Λιβύα ακριβώς τονίζει και καταδεικνύει την ανάγκη να υπάρχει αυτή η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το 2015, όπως γνωρίζετε, οπότε και ξεκίνησε η επιχείρηση με βασική εντολή να προστατευθούν οι ζωέ των μεταναστών με καταπολέμηση του διεθνού εγκλήματο που είναι υπεύθυνο για την διακίνηση αυτών των ανθρώπων. Αυτή ήταν η βασική εντολή. Έκτοτε έχει επιμηκυνθεί και επεκταθεί εντολή καλύπτοντα και την εφαρμογή του ψηφίσματο περί εμπάργου όπλων του Συμβουλίου Ασφάλεια των Αθηνών, καταπολέμηση πετρελαίου, της διακίνησης, παράνομη διακίνησης πετρελαίου, αθρεμπόριο πετρελαίου, και αυτό ε, μέρος της νέας εντολής. Το πρώτο στοιχείο της εντολής, πολέμηση του οργανωμένου κλίματος που για την διακίνηση μεταναστών. Έχουν μειωθεί σημαντικά οι διακινήσεις μέσω της κεντρικής Μεσογείου. Από το 2016 που ήταν η αιχμής. τώρα έχουμε υποχωρήσει ε, κατά 94% σε σχέση με το περσινό έτος. Μόλις 400 μετανάστες πέρασαν μέσω οργανωμένου εγκλήματος. 23.000 ήταν ε, πέρυσι. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στην επιχείρηση Σοφία, που όμως έχει συνεισφέρει σημαντικά και αυτή για την αποφυγή της ε, διακίνησης μεταναστών. Όμως σίγουρα πρόκειται για μια πολύπλοκη πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση με συμμετοχή των χωρών καταγωγής και διέλευσης και επίσης το περισσότερο με την ύπατη αρμοστή για τους πρόσφυγες και το Διεθνή Οργανισμό για τη Μετανάστευση για να μην υπάρξουν καταχρήσεις και παραβίαση των δικαιωμάτων των μεταναστών και στην ίδια τη Λιβύη. Να μην έχουμε πλέον στρατόπεδα κράτησης και να μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί εκτός Λιβύης το συντομότερο δυνατόν. Μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Ένωση με διαφορετικά ε, προγράμματα έχει δώσει βοήθεια για την επιστροφή 43.000 μεταναστών και από τη Λιβύη και έχουν κενωθεί πάνω από 3.300 ε, πρόσφυγες οι οποίοι μετεγκαθίστανται μέσω των προγραμμάτων παροχής βοήθειας και με την ε, συνεργασία όπως είπαμε η Πατιαρμοστία και Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευση. Πολύπλοκη διαδικασία πάντω και σε ό,τι αφορά αυτό το επιχειρησιακό μοντέλο του οργανωμένου εγκλήματο που διακινεί πρόσφυγε και επιχείρηση Σοφία έχει ε, επίσης μια πολύ σημαντική ε, συνεισφορά. Τώρα, άμεσε επιχειρήσεις, διαθαλάσσει και επίσης μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση έρευνες ε, διάσωσης, ε, έρευνες διάσωση, ε, κέντρα συντονισμού, συνεργασία με τη Λιβική Ακτοφυλακή. Ιδίω εντό των χωρικών υδάτων. Εκεί χάνονται οι περισσότερες ζωές, στα χωρικά λιβικά ύδατα. Άρα πρέπει να βοηθηθεί και η λιβική ακτοφυλακή για να σώσει ζωές, ζωές μεταναστών. Η επιχείρηση δεν έχει εντολή ε, για επιχειρήσεις διάσωσης ε, μεταναστών. Πρέπει αυτό να γίνεται σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο. 43.000 νομίζω είναι, πάνω από 40.000 τέλο πάντων, ζωές έχουν σωθεί τα τελευταία χρόνια. Εντολή. Ανανέωση της εντολής. Αυτό αποφασίστηκε στις 26 Μαρτίου επεκτείνεται για μία περίοδο 6 μηνών. Γιατί. Α, και πρόκειται για την ίδια εντολή. Δεν έχει αλλάξει. Με τις τρεις αυτές γραμμές δράσης που σας προνέφερα. Το Συμβούλιο όμως συμφώνησε επίσης παροδικά να μην αναπτύσσονται θαλάσσιες μέσα. Γιατί αυτό. Κατά βάση, διότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συμφωνία ακριβώ πάνω στο πώς οι αποβιβάσεις αυτών δηλαδή που έχουν διασώσει τα σκάφη της Σοφία. Με βάση την αρχική εντολή της επιχείρησης, οι αποβιβάσει όλες θα γίνονταν στα Ιταλικά λιμάνια. Η Ιταλία ήδη από πέρυσι ανακοίνωσε ότι δεν είναι δετεθειμένη να δεχθεί συνέχιση της επιχείρησης από αυτές τις συνθήκες από τον Αύγουστο, είπατε εκπρόσωπο ε, παρουσιάζει στα κράτη-μέλη διάφορες εναλλακτικές προκειμένου να υπερπηδηθεί η δυσκολία αυτή. Δυστυχώς όμως δεν έχει υπάρξει τελική συμφωνία για το χειρισμό αυτού του ζητήματο δεν έχει να κάνει με την εντολή τη επιχείρηση, αλλά αν κάποιο είναι στη θάλασσα, σίγουρα πρέπει να ξέρει τι θα κάνει με τα άτομα που διασώζει σύμφωνα με το διεθνέ δίκαιο και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συμφωνία. Θα ανανεωθεί λοιπόν όπως αποφάσισαν τα κράτη-μέλη η εντολή αλλά θα ανασταλεί η, θαλάσσια, η χρήση θαλάσσιων μέσων. Επίσης μια άλλη απόφαση για να μετριαστούν αρνητικές επιπτώσεις είναι ότι θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί ε, η επιτήρηση από αέρος. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για τις θαλάσσιες επιχειρήσεις. Ενισχύεται λοιπόν η από αέρος επιτήρηση και θα υπάρξει μεγαλύτερη παρακολούθηση και έλεγχος και χερσαία εκ μέρους της ακτοφυλακής που οι άντρε εκπαιδεύονται από την επιχείρηση Σοφία. Επίσης, ξεκάθαρα αναφέρεται στην εντολή ότι το πίεση η Επιτροπή Πολιτικής Ασφάλειας μπορεί να αναθεωρήσει, αναθεωρήσει την απόφασή της και να δώσει περαιτέρω οδηγίες στο διοικητή υπό το πρίσμα διαφορετικής κατάστασης. Αυτή η αναστολή έχει μια σημαντική συνέπεια. Τα κράτη-μέλη, δηλαδή, θα πρέπει να ορίσουν μέσα τα οποία θα μπορούσαν να αναπτυχθούν σε δίποτε χρονική στιγμή αν ε, η Επιτροπή αυτή στο πλαίσιο του Συμβουλίου ή το Συμβούλιο συμφωνήσει ως προς αυτό. Προκαθορισμός δηλαδή των μέσων που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν. Αυτό απαιτείται. Νομίζω αυτά έχω να πω σε σχέση με το που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Θα σταματήσω εδώ την αρχική μου παρουσίαση, αλλά θα σας δώσω ευχαρίστως ε, οποιαδήποτε διευκρίνηση επιθυμείτε. Ευχαριστώ. Okay, Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε και πάλι μαζί μας ε, και που μας αφαιρίζετε τον χρόνο αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. και σας ευχαριστώ που μου δώσω, μας δώσατε και το που βρισκόμαστε. Να ξεκινήσουμε με τους συναδέλφους και με τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί ως τώρα. Θέλετε να έρθετε σε επαφή και με την Προεδρία σε ό,τι αφορά την ε, επιχείρηση Σοφία. Το θέμα της μη ανάπτυξης ε, σκαφών Μας είπατε πόσα άτομα έχουν διασωθεί και για διάφορα ζητήματα. Το θέμα λοιπόν είναι να υπάρξει υποκατάσταση και των άλλων επιχειρήσεων. Αυτό που όλοι διερωτώμαστε είναι το εξή. Αν αφαιρέσουμε τις, α, ε, τους πόρους που δεν θέλουμε να χρησιμοποιούμε και τους αντικαταστήσουμε με δικούς μας πόρους. Το προφανές ερώτημα είναι ότι τελικά θα καταλήξουν να χαθούν ζωές. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό και σε ό,τι αφορά τη Λιβύη και την Τρίπολη. Ε, το ερώτημα και πάλι μπορεί να είναι αφελές, αλλά η υπηρεσία εξωτερικής δράσης πώς αντιμετωπίζει το θέμα της ε, μεταφοράς στην Τρίπολη δεν θα σημαίνει αυτό ότι όλο και πιο πολλά άτομα θα βγουν από εκεί. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό. Δεν θα δημιουργηθεί μεγαλύτερη πίεση και στην περίπτωση αυτή πώς θα διαχειριστούμε και την ανθρωπιστική κατάσταση αλλά και σε ό,τι αφορά την ακτοφυλακή και σε ό,τι αφορά την πολιτική κατάσταση. Είναι ευαίσθητη η στιγμή και μπορεί να τύχει κατάχρηση από διαφόρους για διαφορετικές σκοπιμότητες. Έχετε πολιτική άποψη γι' αυτό. Η κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θυμάμαι ακόμα όταν ε, διώξανε τον Καντάφη και πολλοί Αφρικανοί ε, πιέστηκαν να ανέβουν σε σκάφη για να ε, φύγουν διαθαλάσσεις. Δεν θα έλεγα ότι ανέβηκαν εκεί ο θελός στα σκάφη, τους έσπρωξαν και υπήρξε χαμός και σύγχυση. Τώρα στην Τρίπολη βλέπουμε πολλούς ε, που είναι εσωτερικώς εκτοπισμένοι, όχι αναγκαστικά μετανάστες, αλλά Λίβιους οι οποίοι χρειάζονται ασφαλή λιμένα. Από τις χειρότερες στιγμές όχι απλώς να μην σταματήσει η επιχείρηση Σοφία, αλλά να αλλάξει εντολή και να μην υπάρχουν εκεί καν σκάφη. Ξέρουμε ότι η εντολή είναι η ίδια και έχει αλλάξει ο εξοπλισμός. Μήπως συμβεί λοιπόν τίποτα ανάλογο με το 2011, όπου ο κόσμος ε, διωκόταν, ε, εξαναγκαζόταν να ανέβει στα σκάφη. Οι Αφρικανοί μετανάστες αντιμετωπίζονταν ως φόρη του Καντάφη και αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τη χώρα. Ποιος είναι λοιπόν ο κίνδυνος για τους Λίβιους πολίτες που αναγκάστηκαν να διαφύγουν. Καταλαβαίνω ότι επίσης θα υπάρχουν και αρεοσκάφη στα πλαίσια της επιχείρησης Σοφία που θα κοιτάνε αν υπάρχουν σκάφη που ε, βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση και άνθρωποι που πρέπει να διασωθούν. Οπότε θα αποστέλλονται ανάλογες πληροφορίες στα κέντρα στην Τρίπολη και η τωρινή ε, το φυλακή της Λιβύης, ό,τι και αν γίνει με τον Χαφτάρ, ό,τι και αν γίνει τώρα, θα βοηθηθεί, θα ειδοποιείται να σώζει κόσμο στη θάλασσα. Κόσμο που μπορεί απλώς να διαφεύγει από τις συνθήκες πολέμου για τις οποίες αρχικά, αρχικά μπήκε στη θάλασσα. Να δούμε λοιπόν τι ακριβώς θα κάνουμε. Βοηθούμε την Λιβική Εκτοφυλακή να φέρει κόσμο πίσω στις ακτές και στα κέντρα κράτησης. Αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα. Ή μπορεί να δημιουργήσουμε χειρότερες ακόμα συνθήκες. Να βοηθούμε Λίβιους ε, ταραξίες, όσους είναι κατά του Χάφταρ. Μήπως να διασώζουμε τελικά αυτούς που δημιουργούν όλη αυτή την ε, κατάσταση και την αναταραχή και τους πηγαίνουμε πίσω στην ξηρά. Μήπω είναι η στιγμή τα κάτι μέλη να ξανασκεφτούν τι συμβαίνει, διότι αν αρχίσει πάλι εμφύλιο ή υποδαβλιστή, θα ήταν από τι δυσκολότερε στιγμέ για να αφαιρέσουμε εμεί την παρουσία μας την ναυτική γύρω από τη Λιβύη. Ο κύριος Κώστερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον ε, κύριο Σεράνο για την παρουσίαση της κατάστασης. Είναι σημαντικό ε, να παρατηρήσουμε ότι με την ε, ιδιωτικοποίηση των ε, ε, οργανώσεων έρευνας και διάσωσης και με την αναστολή των επιχειρήσεων ουσιαστικά της Σοφίας δεν υπάρχει πλέον διάσωση διαθαλάσσης και υπάρχει πραγματικά κίνδυνος να υπάρξει κλιμάκωση της κατάστασης και επιδίνωση με απώλειες πολλών ζωών στην Μεσόγειο. και λέει μάλιστα μία αναφορά ότι υπήρχε ένα πιστοποιητικό ε, κάποιων ε, σπουδών ε, που ήθελε κάποιος που πνίκε να το κρύψει αυτό. Ε, Εμεί ως Ευρώπη ε, έχουμε τελικά τον Όρμπαν, τον Σαλβίνη και, τον, ε, και άλλους τέτοιους και ενώ παλιότερα αυτό που μας χαρακτήριζε ήταν ο Βολτέρος και άλλοι διαφωτιστές Έχουμε επιτήρηση ε, από αέρος, έχουμε την ε, Λιβική ακτοφυλακή η οποία επιχειρεί. Δεν ξέρω η ερώτηση και πώς θα απαντηθεί βέβαια. Τι ε, κάνουν αυτά τα αεροσκάφη όταν βλέπουν έναν άνθρωπο μέσα στη θάλασσα. Τους αφήνουν να πληγούν αυτούς τους ανθρώπους, ναι ή όχι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης, ε, τι γίνεται, αυτοί που πάνε να τους βοηθήσουν ε, ουσιαστικά κατηγορούνται ως ε, εγκληματίες και καταδικάζονται γιατί προσπάθησαν να σώσουν 12 χρόνια παιδιά. Τι θα κάνουμε λοιπόν ε, και με τις ε, ενέργειες ε, της Λιβικής Ακτοφυλακής όταν δεν τηρούνται οι διατάξεις του διεθνούς δικαίου. Εσείς ποια άποψη έχετε κύριε Σεράνο. Ναι, είναι ευκαιρία που συζητάμε εδώ την επιχειρήση Σοφία. Διότι θα είναι από τα πρώτα ζητήματα που θα με απασχολούν και στα μέσα μαζική ενημέρωση η Λιβύη και εκτοφυλακή και τώρα με την ε, κατάσταση στην Τρίπολη. Θα παίρνει όλο και μεγαλύτερη δημοσιότητα το θέμα. Οπότε, ο χρόνος περνάει. Ε, πρέπει να το δούμε με μεγάλη προσοχή αυτό. Είναι στο επίκεντρο της προσοχής μας, η κυρία Σπινέλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. ήθελα να εκφράσω την βαθιά μου ανησυχία για την αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής της αποστολής αυτής, της επιχείρησης Σοφία. Η απομάκρυνση των σκαφών, τη στιγμή αυτή και αφού ε, ε, επιδίθηκαν ευθύνε στι ε, μη κυβερνητικέ οργανώσει των ανθρωπιστικών δικαιωμάτων, είναι ένα μήνυμα πολύ σαφέ. Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι ότι η Μεσόγειος θάλασσα αφήνεται τελείως εγκαταλελειμμένη από επιχειρήσεις διάσωσης και ανατίθενται αυτές σε μια Λιβύη που είναι ανύπαρκτη. Δεν υπάρχει Λιβύη ως κράτος. Είναι μια πλάνη, είναι ένα φάσμα. Και είναι και αυταπάτη να νομίζουμε ότι οι ζωές όλων αυτών των ανθρώπων στη Μεσόγειο μπορεί να ανατεθούν ως ευθύνη στα χέρια της Λιβυκής Ακτοφυλακής. Έχουμε αλλάξει τελείως τους όρους του θέματος και πριν από αυτές τις πρώτες επιχειρήσεις και τις αντεπεραθέσει μεταξύ του Χαφτάρ και των αντιπάλων του. Είναι λοιπόν κάτι που μας ανησυχεί βαθιά. Κατά την άποψή μου πρέπει να το ξανασκεφτούμε, διότι δίνουμε την εντύπωση ότι υπάρχει μια περίεργη ισορροπία τρόμου στη Μεσόγειο. Δηλαδή η αποτροπή ουσιαστικά το αποτρεπτικό στοιχείο είναι ο θάνατος των μεταναστών. Δηλαδή, εάν πεθάνουν μετανάστες, έχει επιτευχθεί ο τελικός σκοπός και η λύση. Είναι σοβαρότατο και θυμίζω ότι και ο Πάπας αυτό ακριβώς είπε. Το να μην βοηθούμε τους ναυαγούς, το να αφήνουμε τους ανθρώπους να πνίγονται, τι είναι αυτή, είναι επιλογή της Ευρώπης, το είπε ο ίδιος ο Ποντίφικας. Και ένα δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η απαρχή της απόφασης αυτής για τον εξοπλισμό της Λιβικής Ακτοφυλακής έχει να κάνει με το ότι η Λιβύη θεωρείται ε, ασφαλής χώρα για αποβίβαση. Ακόμα και αν πείτε ότι δεν είναι ασφαλής τώρα, εφόσον εξαπλίζεται τη Λιβύη Ακτοφυλακή, να λες και τη θεωρείται τέτοια. Ε, πριν από δύο χρόνια ο ΙΕ έλεγε ότι δεν είναι ασφαλής χώρα. Τις προηγούμενες μέρες εν μέσω πολέμου του Χάφταρ και του Σαράζ, ο κύριος Γκουτιέρες, ο γενικός γραμματέας του ΙΕ, επισκέφθηκε, επισκέφθηκε ένα καταβλισμό προσφύγων, κράτησης ε, μεταναστών στην Τρίπολη και είπε ότι ήταν deeply shocked, ότι συγκλονίστηκε και κανείς δεν μπορεί να πει σε αυτή τη φάση ότι η Λιβύη είναι ασφαλής λιμένας για αποβίβαση δήλωσε. Αυτοί οι καταβλισμοί ε, προσφύγων δεν είναι μόνο ευθύνη της Λιβύης. Είναι ευθύνη ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας. Αυτό το είχε πει ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΤΟΥΙΕ. Και τώρα το δικό μας το σχέδιο θα πούμε ότι λειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Και αυτό που πρέπει να πω οπωσδήποτε είναι ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα κέντρα κράτηση, στου καταβλισμού δηλαδή, είναι κάτι που πρέπει να το δούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Στον καταβλισμό τη Τρίπολη, οι κρατούμενοι αναγκάζονται να βγουν από τα κελιά και τους πετάνε στα χέρια όπλα και τους στέλνουν να πολεμήσουν τον Χαφτάρ και φωνάζουν οι κρατούμενοι ότι θέλουν να επιστρέψουν στα κελιά τους Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Είναι φρικαλαίο. Μιλάμε για ρεπορτάζ το οποίο προβλήθηκε πάρα πολύ ε, στους Irish Times από την κυρία Χάιντεν και επ' αυτού ε, εξαιτίας αυτών των ειδήσεων για το πώς ε, χειραγωγούνται οι κρατούμενοι, πως του αναγκάζουν να πάρουν μέρο στον πόλεμο. Γι' αυτό ξεκίνησε να κάνει αυτέ τι δηλώσει ο Κουτιέρε. κάνει όλη την επίσκεψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Μπάρμπαρα. Συνάδελφοι, λίγο έχασα την αίσθηση του χρόνου και έχουμε ψηφοφορίες στι 4.30. Η κυρία Γκόμες και εγώ μακρηγόρησα, δεν λέω, αλλά σα παρακαλώ ένα λεπτό καθένα για να προλάβουμε να έχουμε και κάποιε απαντήσει. Ναι, με συγχωρείτε, Αλλά ένα λεπτό όλοι σα για να προλάβουμε να ακούσουμε και τι απαντήσει. Μπίργκιτ, πρώτη, μετά η Άννα και μετά η Μαίτε. Ευχαριστώ πολύ και νομίζω ότι θα είμαι και πολύ σύντομη. Πολλά τα ακούσαμε ήδη. Αλλά ανησυχώ λίγο γιατί μιλάμε πάρα πολύ εδώ αυτές τις ημέρες για την ε, παραπληροφόρηση και μήπως ε, σήμερα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για παραπληροφόρηση ή να μας δημιουργήσει έκπληση οι δημιουργικέ εκφράσει που έχουν χρησιμοποιηθεί. Καταρχάς λοιπόν μιλάμε ότι η δραστηριότητα, η επιχειρήση Σοφία συνεχίζεται. Εγώ δεν βλέπω να συνεχίζεται. Είναι διαφορετικό να παρακολουθούμε την κατάσταση από αέρος. Είπατε ότι οι πιο πολλοί μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στη Λιβική θάλασσα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ε, σώζουμε ζωές. Δεν, δεν σώζουμε ζωές. Ξέρουμε τι συμβαίνει στη Λιβύη και ξέρουμε τι παθαίνουν οι μετανάστες. Ε, περνάνε από βασανιστήρια, σκλαβιά. Δεν βλέπω να σώζουμε ζωές. Και δεν είμαι βέβαιη κατά πόσο μπορούμε να το αποκαλέσουμε αυτό κατά χρήση του μεταναστών στη Λιβύη. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έκφραση. Όταν μιλάτε για οργανωμένο έγκλημα, ότι φεύγουν οι μετανάστες δηλαδή από τις ακτές αυτές και έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα τι άλλο τρόπο έχουν αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται σε έσχατη ανάγκη προστασίας. Μιλάμε για επανεγκατάσταση. Εγώ δεν βλέπω αριθμητικά στοιχεία εύλογα για να δικαιολογήσουν όλα αυτά. Αναρωτιέμαι λοιπόν πραγματικά αν θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε χρησιμοποιώντας αυτές τις εξηγήσει. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Η κυρία Κόμες, καλώς όρισατε κυρία Σεράνο. Γιατί έληφθη αυτή η απόφαση να σταματήσουν ε, οι χρήση πλοίων Αυτό σημαίνει ότι θα καλέσει η κυβέρνηση της ΜΚΟ να, σώσουν τις ζωές πέρα από τα, τους πόρους αυτούς ε, αντί να τους ε, κατηγορούμε να λέει η Επιτροπή ότι η ΜΚΟ δεν θα πρέπει να ποινικοποιούνται, θα πρέπει να απαγορεύεται αυτό. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν, ότι ζητάμε πλέον από τις ΜΚΟ να κάνουν και να αντικαταστήσουν ε, την επιχείρηση Σοφία. Και η επίθεση Μπαφτάρου ουσιαστικά θέλει να διασπάσει την ε, συνοχή της κυβέρνησης. Τι βλέπουμε λοιπόν, ότι όχι μόνο οι περιφερειακές δυνάμεις και το παιχνίδι των δυνάμεων που περιλαμβάνει το Κατάρ και την Αίγυπτο Και τι γίνεται και στα κράτη-μέλη. Πού είναι το κράτος δικαίου. Όλοι βλέπουμε πίσω από τη Σαουδική ε, Αραβία και την Αίγυπτο να κρύβονται. Θα κάνουμε τα ίδια ακριβώς σφάλματα του παρελθόντος. Πριν του κατάφυγε. ναι. Διακόπτει ο Πρόεδρος. είτε ένα λεπτό. Δεν θέλω να καθυστερήσουμε δύο λόγια να πω μόνο. Το πρώτο, πολύ λένε ότι ε, εκτελούν εντολές και δεύτερον αντιμετωπίζουμε ανθρώπους σαν ζώα. Thank you very much, Maite. Ευχαριστώ, Μαϊτά. Σε ευχαριστώ γιατί ήσουν και συντομή. Και εύστοχη. Προφανώς το θέμα λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ επίμαχο. Για πείτε μας λοιπόν έχετε να μας απαντήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καταλαβαίνω ότι είστε ανακανακτισμένοι και, ε, και εμείς ε, συμμεριζόμαστε την αγανάκτηση αυτή. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Και ασφαλώς πιστεύω ότι όλοι όσοι βλέπουν τι σημαίνει στη Λιβύη είναι αγανακτισμένοι, εξοργισμένοι μάλιστα λόγω του τι συμβαίνει, λόγω του κινδύνου για τις ανθρώπινες ζωές. Αυτό δεν χωράει αμφιβολία και δεν νομίζω ότι είναι κανείς που να λέει ότι βρισκόμαστε σε καλή κατάσταση. Ωστόσο, έχω να πω, η απόφαση που ελήφθη για την παράταση της εντολής ελήφθη πριν, πριν από τις κινήσεις αυτές. Δεν είχε συναπολογιστεί λοιπόν στη λήψη της απόφασης. Επίσης να πω ότι η απόφαση που ελευθεί προβλέπει την δυνατότητα ανάπτυξης δυνάμεων εκ νέου αν αυτό χρειαστεί. Όπως σας είπα στην αρχή, η αναστολή δεν σημαίνει ότι αν χρειαστεί δεν θα είναι στη διάθεσή μας η πόρη αυτή θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο ρόλος και η εντολή της επιχείρησης Σοφίας ήταν να διασωθούν ζωές μέσω της καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Δεν ήταν ε, λοιπόν γενικά και αόριστα η διάσωση ανθρώπων. Φυσικά και θα πρέπει να διασωθούν άνθρωποι, αλλά ακόμα και αριθμητικά η επιχείρηση Σοφία έχει καλύψει πάνω από το 1 πέμπτο των διασώσεων. και υπάρχει ευθύνη διάσωσης από το Ναυτικό Κέντρο Συντονισμού. Κάποιοι ρώτησαν τι κάνουν ε, οι δυνάμεις μας όταν ε, εντοπίζουν ε, άτομα σε κίνδυνο. Επικοινωνούν με το Ναυτιλιακό Κέντρο Συντονισμού. Και ο συντονισμό είναι λοιπόν δική του αρμόδιότητα. Είτε μα αρέσει είτε όχι. Στην πραγματικότητα, τα σκάφη των μεταναστών και όπως ξέρετε από τις τελευταίες εξελίξεις, ε, πολλοί μετανάστες ε, βρίσκονται σε, σε πιο κάρεβα και δεν μπορούν να ξεπεράσουν ε, τα όρια των τοπικών χωρικών υδάτων. Η επιχείρηση Σοφία, λοιπόν, αυτό που κάνει και με άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να εκπαιδεύει τη Λιβυϊκή Ακτοφυλακή προκειμένου να μεταχειρίζεται τους ανθρώπους αυτούς με τον πιο ανθρώπινο τρόπο. Δεν ε, δικαιολογούμε το πώς ε, μεταχειρίζονται τους μετανάστες στη Λιβύη. Εδώ δεν χωράει αμφιβολία και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ξεκάθαρη και υπάρχει συνεργασία και με τον ΟΗΕ με σκοπό να αλλάξουν ακριβώ οι συνθήκες διαβίωσης και μεταχειρίσης των ανθρώπων αυτών. Η κατάσταση στη Λιβύη λοιπόν είναι αυτή που γνωρίζετε. Δεν νομίζω ότι οποιοδήποτε είναι ικανοποιημένο με αυτό που υπήρχε και πριν από την επίθεση, ούτε με την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε τώρα. Και ναι, είναι σημαντικό να βρούμε μια βιώσιμη λύση και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να δράσουμε πιο αποτελεσματικά και να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά τα θέματα μεταναστών. και, και θα προκαλέσει αυτό πιο πολλά προβλήματα. Δεν ξέρουμε, είναι δύσκολο να το προδιαγράψουμε. Θα υπάρχουν πιο πολλές μετακινήσεις. Θα είμαστε έτοιμοι όμως να αντιδράσουμε. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι αυτό δεν αποτελεί λύση. Και δεν είναι ικανοποιητική λύση. Και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά την κατάσταση. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των ατόμων που πλήττονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σεράνο, λέει ο Πρόεδρος. αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει με κάποιον πιο υψηλό εξωματούχο και από την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα. Ε, δεν είναι εδώ η Προεδρία. γιατί νομίζω ότι έτσι μπόρεσαν ε, οι βουλευτές της Επιτροπής να μεταφέρουν τα σημαντικά μηνύματα που είχαν κατά νου σε ό,τι αφορά τη Λιβύη. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τι ερωτήσει αυτέ και τις απαντήσεις που δώσατε στις ερωτήσει Προφανώς και η κατάσταση προκαλεί αγανάκταση, αλλά νομίζω ότι μα δώσατε απαντήσεις και αυτό είναι σημαντικό. Συνάδελφοι, θα ψηφίσουμε σε ένα λεπτάκι. Ελικονικά, Αν υπάρχουν ε, αναπληρωματικοί, θα ξεκινήσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Συνάδελφοι, αν είσαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Να διαβάσω μία εισαγωγή για την πρώτη ψηφοφορία. Παρακαλώ, διακαθίστε λοιπόν. Να περάσουμε στην πρώτη ηλεκτρονική ψηφοφορία, στο σημείο 6, η πρόταση για φαρμαστοπική απόφαση για την απόφαση της Eurojust για τη Σύμφωνια Δικαστικής Συνεργασίας σε ποινικά θέματα μεταξύ Eurojust και του Βασιλείου της Δανίας. Τα γνωρίζετε οι συνάδελφοι επειδή δεν υπήρξε ψηφοφορία, ε, μάλλον συζήτηση. Να σας διαβάσω τι ψηφίζουμε αν ε, έχετε λίγο μονή, να σας διαβάσω. Απλοποιημένη διαδικασία επιβεβαιώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από την Επιτροπή μέσω για την διαβούλευση να ολοκληρωθεί πριν από τέλο τη θητεία και ω ε, πρόεδρο τη ΛΥΜΠΕ, η Eurojust, η Δανία, η Επιτροπή και η Προεδρία παρουσίασαν την προστασία αυτή την προηγούμενη εβδομάδα στι 2 Απριλίου και όλε. Ε, οι πλευρέ ε, ευχαριστούν το Κοινοβούλιο που επιτάχυνε τι διαδικασίε. Το σχέδιο απόφαση και η συμφωνία σα απεστάλησαν. Πρόκειται για μια διαδικασία μέσω διαβούλευση, όπου εκφράζουμε τη γνωμοδότησή μα για μέχρι σε ένα συγκεκριμένη προθεσμία. Αποφασίσαμε λοιπόν το εξή: συνεχισμό στη συνέχιση τη ε, ε, συμμετοχή τη Δανία στη Eurojust για τη χρηματοδότηση της Eurojust το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη, συμμετοχή στη Σέγγεν και δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων και τέλος εφαρμογή του EDPS και ίσχυν τα δικαιώματα του δικαστηρίου του Ευρωπαϊκού Κοινοτήτων. Συνεπώ, όσοι εισηγητή, ε, προτείνω την επιβεβαίωση της απόφαση αυτή και καλό παράλληλα τις πολιτικές ομάδες να προσταθεί το θέμα αυτό στην ε, τελευταία ολομέλεια προς ψήφιση και έτσι λοιπόν μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Εάν ψηφίσατε όλοι σας, άμα. Πέρας ψηφοφορίας. 37 ψήφοι υπέρ, καμία κατά, μία αποχή. Άλλη μία ψηφοφορία είχαμε η οποία αναβλήθηκε, το 7, με ψηφοφορία για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας. Περνάμε λοιπόν στο 8 πρόληψη του, της διάδοσης υλικού τρομοκρατικού στο διαδίκτυο. Και τώρα μιλάμε λοιπόν ε, για την γνωμοδότηση. Ο κύριος Ντάλτον είναι ο εισηγητής. Ο κύριος ε, Ντάλτον θέλει να πάρει το λόγο σε ό,τι αφορά την έκθεση πρόληψη τη διάδοση του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Θέλετε να πάρετε το λόγο, κύριε Ντάλτον. Ναι, ναι. Το μικρόφωνο μου είχε ένα πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα μόνο να επισημάνω κάποια στοιχεία, αν μου το επιτρέπετε. Να ευχαριστήσω καταρχά όλου του συναδέλφου για τη δουλειά που έκαναν και προσπάθησαν να βελτιώσουν το κείμενο αυτό τη Επιτροπή. Να πω ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει χώρο στο διαδίκτυο για τρομοκρατικό περιεχόμενο. Ωστόσο, ο συμβιβασμό παίρνει καιρό ε, έχουμε περίπλοκα ζητήματα μπροστά μα και μα ανησυχούν κάποια ζητήματα και οι βουλευτέ θα πρέπει να τα κοιτάξουν όλα αυτά με προσοχή. Το κάναμε λοιπόν αυτό από κοινού. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να πιστεύει ότι οποιοδήποτε θέλει να αλλάξει μία πρόταση χρονοτρεβεί ή τα παίρνει από την Google και από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό το βλέπουμε λοιπόν σε πολλές περιπτώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το είδαμε και για το copyright και αυτό καταδεικνύει ότι δεν υπάρχει σεβασμό για το Κοινοβούλιο και κατανόηση για τα μέλη του Κοινοβουλίου. Δεν ληστεύει αυτό, δεν στέκει. Και υπάρχει λοιπόν μια συκοπατική ε, εκστρατεία κατά του Κοινοβουλίου στις, σε εφημερίδε, οι οποίε θα πρέπει να εξτρακτεί και λίγο παραπάνω. Δεν είναι λοιπόν ε, δική μας δουλειά να σκεφτόμαστε το κλειδοβότημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δουλειά μας είναι να εξετάσουμε ένα πολύ σύνθετο νομοθέτημα και αυτό το κάνουμε λοιπόν τους τελευταίους μήνες. Και θα ήθελα να σας πω λοιπόν το χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο εργαστήκαμε για να μην υπάρχει καμία ψευδέστηση για το πόσο γρήγορα δράσαμε. Η Επιτροπή μας ε, πήρε μέσα Ιανουαρίου αυτή την πρόταση μόλις ε, καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα που είχαμε. Μόνο λίγε μέρες αργότερα ήταν έτοιμη η έκθεσή μου και το ψηφίζουμε τώρα λοιπόν αυτό στις 10 Απριλίου 8 Απριλίου με δύο μικρές καθυστερήσεις. Αυτή είναι η σωστή κοινοβουλευτική διαδικασία. Να είμαι λοιπόν σαφέστατος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι κάναμε σωστά τη δουλειά μας. Κανείς δεν τα παίρνει από μεγάλες επιχειρήσεις και σας παρακαλώ στο μέλλον να σέβεστε τις ε, διαδικασίες, τις κοινοβουλευτικές ε, δουλέψαμε σκληρά και θεωρώ ότι πετύχαμε ένα καλό νομοθέτημα και ελπίζω μετά τη σημερινή ψηφοφορία να έχουμε μια ισχυρή εντολή του Κοινοβουλίου για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον εισηγητή, λέει ο πρόεδρος, αγαπητοί συνάδελφοι. Προφανώς το θέμα αυτό είναι λίγο περίπλοκο και η ψηφοφορία είναι λίγο περίπλοκη. Σας παρακαλώ να επιδείξετε ψυχραιμία και υπομονή για να την ολοκληρώσουμε. Θα σας λέω λοιπόν τη σελίδα που θα βρίσκομαι στην ε, δικό μου κατάλογο, μπορεί να είναι διαφορετικός από το δικό σας. Συμβαστική 1. Όλα ηλεκτρονικά παρακαλώ. Να κοιτάξουμε αν είσαστε όλοι παρόντες και αν είσαστε όλοι στις θέσεις σας. Κάποιοι ψήφισαν ήδη. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Λίγα δεύτερα ακόμα. Μέχρι ότου καθίσατε τα ψήφισατε, παρακαλώ όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην σελίδα 40 στη δική μου ε, αριθμίση που είναι ο συμβιβασμός υπαριθμών 2. Συμβιβασμός υπαριθμών 2. υπομονή για να μην κάνουμε λάθη. Αν ψηφίσατε όλοι, συμβαστική 2. Ψηφίζουμε. Αν ψηφίσατε όλοι σας, ε, πέρασε. Εγκρίνεται. Σελίδα 30 τώρα. Αντιλογική σκέψη 9 λογική σκέψη 9. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Η 89, τροπολογία 89, ναι, μπράβο Μπρίκετ. Σωστά τα λες. Εάν ψήφισατε όλοι παρακαλώ πέρα ψηφοφορία. Εγκριθήκε. Συμβαστική 3. Σελίδα 31. Συμβαστική 3 παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Σελίδα 34. Συμβιβαστική 4α. Συμβαστική 4α ψηφίζουμε. Η 4α. μου ψηφίσετε παρακαλώ όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4 στην ίδια σελίδα ψηφίζουμε. Συμβαστική 4. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Και τώρα πάμε τη συμβαστική 5. Σελίδα 48. 48 σελίδα. Ψηφίζουμε παρακαλώ για την συμβαστική 5. Αν ψήφισατε όλοι, πέρας. Εγκρίθηκε. Σελίδα 51 τώρα. Συμβαστική 6. Συμβαστική 6. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 7. Σελίδα 68. Η συμβαστική 7. Ψηφίζουμε παρακαλώ τη συμβαστική 7. Εάν ψηφίσατε όλοι σας. Πέρασε. Εγκριθήκε. Συμβαστική 8 στη σελίδα 73. Συμβαστική 8. το παρακαλώ όλοι, πέρας. Εγκρίθηκε. Σελίδα 78, τροπολογία 570. Η 570 λοιπόν στη σελίδα 78. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Συντώ συγγνώμη και δείξτε υπομονή. Είναι από κοινού. Οι 570 με την 146 ψηφίζουμε. ...570 και τον 146. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβαστική εννέα. Συμβιβαστική εννέα, στην ίδια σελίδα παρακαλώ ψηφίζουμε. Πέρας. Σελίδα 81, συμβαστική 10. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 11 στη σελίδα 83. 11 παρακαλώ. Συμβαστική 11. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 12 στην σελίδα 86. Συμβαστική 12 παρακαλώ. ψηφορέας Εγκρίθηκε. Και τώρα πάμε στην σελίδα 88, 613. Η 613 στην ε, σελίδα 89. Αν ψηφίσετε όλοι, πέρα ψηφορίες. Απορρεύθηκε. 611 παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 13. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Πάμε τώρα στη συμβαστική 14, στη σελίδα 93. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε στη σελίδα 95, συμβαστική 15. Συμβαστική 15. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 657. 657 στη σελίδα 97 από κοινού με την μέχρι ότου μαζί με την 660, 657 μαζί με την 660. Και πάμε στην 228 ε, και ΜΚΟ 32. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 16. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 17. Πέρασε. Συγγνώμη, ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 18. Σελίδα 109. Ψηφίζουμε. ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. 715-716 ψηφίζουμε παρακαλώ τώρα τροπολογίες. Πέρας. Εγκρίθηκαν. Καλτ 83, παρακαλώ ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 19. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 20. Ψηφίζουμε. Πέρας. Και αυτό εγκρίθηκε. 726 τροπολογία τώρα. Ψηφίζουμε την 726. Περάς. Εγκρίθηκε. 734 και ΙΜΚΟ 123 είναι ταυτόσιμες. Παρακαλώ ψηφίζουμε. Περάς. Απορρεύτηκε. 732. Ψηφίζουμε. «732, 733 ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε. Εγκρίθηκε. ΙΜΚΟ 129. Στα παραρτήματα. Παρακαλώ ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Αντιλογικές σκέψεις. 48 παρακαλώ. Ψηφίζουμε την τροπολογία 48. Απορρίφθηκε. 49 παρακαλώ ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίφθηκε και περνάμε στην ΚΑΛΤ 3. Ε, Α, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. Ξεχάσαμε την ΕΜΚΟ 2. Ψηφίζουμε την ΕΜΚΟ 2. Πέρας. Εγκρίθηκε. Καλτ 3. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Καλτ 8. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορριφθήκε. Ήμκο 9. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίφθηκε. Ήμκο 10. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίφθηκε. Η 112. Πέρας. Εγκρίθηκε. 113. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίφθηκε. 206. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίφθηκε. 205. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίφθηκε. Κάλτ 21. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίφθηκε. 207. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. 209. Ψηφίζουμε. Πέρας. Η 209. 209. Να ψηφίσετε όλοι σας παρακαλώ. Πέρας. Απορρίφθηκε. Καθυστερήσα λίγο. Να περάσουμε στην 200. 210 παρακαλώ. 210. Ε, Πέρασε. Εγκρίθηκε. Η 211. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Ήμκο 29. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίφθηκε. 216 και 217. Ταυτόσημα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίφθηκε και τελική ψηφοφορία. Α, έχουμε και την 218. 218 παρακαλώ ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορριφθήκε. Και τώρα με μονομαστική κλίση στην τελική ψηφοφορία, στο κείμενο που στροποποιήθηκε. Ψηφίζουμε, παρακαλώ. Το ΕΛΚ καταψηφίζει, δεν, μπορεί, δεν νομίζω. Ψηφίζουμε, παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε 35 ψήφοι υπέρ, μία κατάκτω αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή.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 Συνάδελφοι, έχουμε δύο ακόμη σημεία στην ημερήσια διάταξη για τώρα το απόγευμα. Εάν μείνετε, μείνετε. Αλλιώ φυγέτε. Αλλά ησύχω, παρακαλώ. Uh, Να περάσουμε στο σημείο 10. Ερώτηση που περιμένει γραπτή απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία επέβαλε η Σόφη Ιντφέλτ για τον ε, νόμο προστασία των δεδομένων και την τήρηση δεδομένων χωρίς ε, την συνένεση για τα πολιτικά κόμματα στην Ισπανία. Από τις 27 Φεβρουαρίου έχει τεθεί η ερώτηση και βάσει του άρθρου 103.5 του ιστορικού κανονισμού οι ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν ενώ εντός της προθεσμίας που αυτό το άρθρο ε, συζητιούνται στη συνεδρίαση. Αυτό συμβαίνει λοιπόν εδώ και ε, οι συντονιστές ζήτησαν να απαντηθεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής. Κυρία Ιντβελτ, μπορείτε να συζητήσετε με τον κύριο Μίκολ, Γενικό Διευθυντή από την DigiJust, το θέμα σας. Σόφη, έχετε το λόγο πρώτη. Είναι βεβαίως προφανές, αλλά Παρακαλώ πείτε γιατί ε, θέσατε το ερώτημα και θα περάσουμε στην Επιτροπή. Ε, ναι, ευχαριστώ τον Νοέμβριο. Στα τέλη Νοεμβρίου υποβάλαμε ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ε, Ισπανικό νόμο προστασία των προσωπικών δεδομένων που επιτρέπει στα πολιτικά κόμματα να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των πολιτών χωρίς τη συνένεσή τους. Και αυτό αρχίζει να γίνεται πιεστικό ζήτημα, διότι στην Ισπανία θα γίνουν εκλογές στα τέλη του μήνα. Και στο τέλο του επόμενου μήνα θα έχουμε και τι ευρωεκλογέ. Λάβαμε απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ουσιαστικά λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σμερίζεται τις δικές μας ανησυχίες και θεωρεί ότι η διευκρίνηση από τις ισπανικές αρχές εφόσον δοθεί θα είναι και το, η ένδειξη για το πώς να προχωρήσουμε. Δεν είχαμε όμως καμιά περαιτέρω αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η απάντηση αυτή ε, είναι από τις 28 Φεβρουαρίου. Εν τω μεταξύ, ο νέος νόμος, αυτή η νομοθετική αλλαγή, έχει αποτελέσει αντικείμενο αμφισβήτησης στα ισπανικά δικαστήρια και τα ισπανικά δικαστήρια έχουν δώσει προθεσμία ως τις 2 Απριλίου στην ισπανική κυβέρνηση για να απαντήσει. Ε, κατόπιν τα δικαστήρια θα εξέδεδαν απόφαση εντός δεκαημέρου. Ε, βέβαια εκεί ισχύουν και άλλοι κανόνες, 30 ημέρες σε συγκεκριμένες συνθήκες, αλλά νομίζω τα ισπανικά δικαστήρια θα έχουν ε, κάθε λόγο να δώσουν ε, την απάντησή τους, να εκδώσουν την απόφασή του πριν τις 28 Απριλίου, που είναι οι Ισπανικές εκλογέ και σίγουρα και πριν τι ευρωεκλογέ. Και φαντάζομαι ότι αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα αυτό οι ισπανικέ αρχέ, διότι αυτό που προκύπτει ε, από το τι έχει γίνει ως τώρα είναι ότι το δικαστήριο σε ολομέλεια εξετάζει το θέμα. Δεν ξέρω πώ το λένε αυτό σωστά. Θα ήθελα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα ενημερώσει για την κατάσταση των πραγμάτων. Δεν ξε... μπορεί φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει εκ μέρου τη Ισπανική κυβέρνηση, αλλά το ζήτημα είναι σημαντικό. Διότι όλοι λένε πώ θα βεβαιωθούμε ότι οι εκλογέ είναι ελεύθερε, ανεξάρτητε, δημοκρατικέ, ότι δεν υπάρχει περί παρεμβολή. Πριν από ένα χρόνο όλοι σοκαριστήκαμε με τις αποκαλύψεις για, το, για την Cambridge Analytica και πώς χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα για την ε, νοθεία ή τέλο πάντων τη χειραγώγηση στις εκλογές. Είναι λοιπόν αρκετά ε, φοβερό να προβλέπουν τέτοιου νόμου οι κυβερνήσει ε, των ευρωπαϊκών κρατών. Είναι ε, τελείω αντίθετο με όσα συζητάγαμε και νομοθετούσαμε τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Τι έχει κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη στιγμή που μα έστειλε την πρώτη τη απάντηση στην στις 28 Φεβρουαρίου. Έχετε κάτι επιπλέον να μας πείτε για την ε, εκδίκαση της υπόθεσης. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και καταρχάς να με συγχωρείτε που στείλαμε αυτή την απάντηση πέραν των προκαθορισμένων προθεσμιών, χίλια συγγνώμη, αλλά πραγματικά αφού ενημερωθήκαμε και λάβαμε και ενημέρωση από το Κοινοβούλιο και από τις Ισπανικές Αρχές για τον Ισπανικό νόμο, αποταθήκαμε στο Ισπανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης. και το συζητήσαμε και με την IEPD, την Ισπανική Αρχή για την Προστασία των Δεδομένων, η οποία με εγκύκλιο έχει ερμηνεύσει το νόμο αυτό για τις ε, διασφαλίσεις που προσφέρονται στην ερμηνεία του άρθρου 28 του Ισπανικού νόμου. Συγκεκριμένα ότι αυτή η αρχή Τη Ισπανία θα πρέπει να δίνει την ε, δική τη άποψη ότι όλα αυτά να γίνονται εντό των πλαισίων του Ισπανικού Συντάγματο και ούτω καθεξής. Όμω όπω ε, είπατε και εσεί, και καθώ ήμασταν και σε συνεννόηση με τι ισπανικέ αρχέ και τον DPA, την αρχή για την προστασία των δεδομένων τη Ισπανία, Περιμένουμε τώρα να εξεταστεί και η προσφυγή από τον Ισπανό διαμεσολαβητή, κάτι που έγινε παραδεκτό από το Ισπανικό δικαστικό σύστημα, τα δικαστήρια. Από τη δική μας λοιπόν την πλευρά η συζήτηση συνεχίζεται με τις εθνικές ε, αρχές με, όλ, με τη συμμετοχή όλων και περιμένουμε το αποτέλεσμα αυτών των ε, δικών, των υποθέσεων. Έχουμε διμερείς ε, συζητήσεις που προβλέπονται στο εγγύς μέλλον με τις Ισπανικές Αρχές και θα το ξαναθέσουμε το θέμα. Σε αυτήν όμως τη φάση Περιμένουμε η υπόθεση να εκδικαστεί στα δικαστήρια. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που η Κομισιόν ε, το πήρε σοβαρά το θέμα για τις επαφή με τις Ισπανικές Αρχές, όμως υπάρχει και θέμα χρόνου εδώ δεν αρκεί το ότι απλά μας λέτε ότι παρακολουθείτε την κατάσταση. Σε τρεις εβδομάδες και λιγότερο από τώρα γίνονται εκλογές στην Ισπανία. Μετά θα πούν ναι υπήρχε πρόβλημα. Μα δεν ε, είναι, αυτό αποδεκτό. Δεν είστε εσείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επόψη των ε, δεδομένων. Όμω πρέπει παρόλα αυτά να επιβλέπετε την εφαρμογή τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και εδώ ο χρόνο είναι χρήμα. Τι θα κάνει η Κομισιόν ώστε τα δεδομένα αυτά να μην χρησιμοποιηθούν για χειραγώγηση των εκλογών. Πώς θα αποφύγετε τον κίνδυνο αυτό πριν τις 28 Απριλίου, όχι κάποια στιγμή στο μέλλον. Χρησιμοποιούνται τα δεδομένα στο πλαίσιο μιας προεκλογικής εκστρατεία που έχει ήδη ξεκινήσει, άρα ήδη γίνεται ζημιά. Τι κάνει λοιπόν κατεπηγόντας η Κομισιόν. Please go ahead. Well. Απαντήστε παρακαλώ. Δύο σκέλη έχουμε εδώ. Πρώτον, να ξεκαθαρίσω ότι το γεγονός ότι γίνεται επεξεργασία άνευ σε εγκαταθέσεως. Αυτό δεν συνιστά παραβίαση τη ομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, γιατί μπορεί η επεξεργασία των δεδομένων στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού να γίνεται για διάφορου λόγου. Και ένα από του λόγου αυτού είναι η εθνική νομοθεσία που παρόλα αυτά προβλέπει, έχει έγκαια ασφαλιστικέ δικλείδε. Η ανησυχία μα τώρα έγκυται στη διατύπωση του άρθρου κατά πόσον παρέχονται όλες οι ασφαλιστικές δικλείδες από την Ισπανική νομοθεσία. τη δική της ερμηνεία η αρμόδια Ισπανική αρχή και λέω ότι παρέχονται όλα τα απαραίτητα εχέγγυα. Εν τω μεταξύ περιμένουμε την έκβαση της δίκης. Υπάρχουν όμως αυτά τα ηχέγγια τα οποία έχει προβλέψει επιπλέον πλέον η Ισπανική Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Που γνωρίζει απολύτως τις ανησυχίες μας, αλλά επειδή είναι σε εξέλιξη δίκη εμείς δεν μπορούμε να αναλάβουμε δράση στο μεταξύ. Πρόεδρος. Θέλετε ξανά το λόγο. Καταρχάς, μια εγκύκλειος είναι ένα επεξηγηματικό φυλάδιο. Δεν είναι νομική διασφάλιση, δεν είναι ένα χέγγιο από νομική πλευρά, δεν έχει το ίδιο καθεστώ, άρα δεν αρκεί. Φυσικά και δεν μπορείτε εσείς να παρέμβετε στη δίκη, αλλά αυτό που μπορείτε να κάνετε με ένα από τα καθήκοντα της Κομισιόν εξασφαλίζει την ορθή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Άρα έχετε αρμοδιότητες, έχετε εξουσίες, όχι στο πλαίσιο αυτής της δίκης, αλλά να πείτε στις Ισπανικές Αρχές ότι εμείς πιστεύουμε πως τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται την νομοθεσία δεν συνάδει με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Γιατί δεν συνιστά νομικό χέγγι αυτή η εγκύκλειος και έχουμε και το στοιχείο του χρόνου, όπως είπα. Εμείς 22 Νοεμβρίου καταθέσαμε το ερώτημα. Έχει περάσει αρκετός καιρός έκτοτε. Γιατί πρέπει να ξαναπεριμένουμε τώρα για να καταλήξουμε λίγο πριν τις εκλογές, το συμπέρασμα ότι ναι, ίσως υπήρξε ε, χρησιμοποίηση αυτών των στοιχείων για χειραγώγηση των εκλογών. Τελευταία απάντηση από την ε, Κομισιόν και θα κλείσουμε. Ναι, ευχαριστώ. έχουμε ανησυχίες με το άρθρο και αυτό το έχουν καταλάβει, το έχουν πάρει το μήνυμα οι Ισπανικές Αρχές. Τους το είπαμε και το κατάλαβαν. Τι άλλο να κάνουμε, υπουργό, ε, ο Επίτροπος έγραψε στον αρμόδιο υπουργό. Δεν μπορούμε να πάμε σε πιο υψηλό επίπεδο. Έχουμε και διμερείς αρχές επαφές και στις ευδημερίες αυτές επαφέ έχουμε μεταφέρει το μήνυμα στις πολιτικές αρχές, σε επίπεδο εργασίας. Το συζητάμε με τις αρχές προστασία δεδομένων. Υπάρχει αυτή η κύκλος που όπως πολύ σωστά λέτε βέβαια δεν είναι νομοθέτη. Αλλά υπάρχει αυτή η ερμηνεία της Ισπανικής Αρχής και εφαρμογή της νομοθεσίας επί τόπου. Αυτά είναι κάποια πρόσθετα εχέγγυα δεν θέλω να ακουστώ γραφειοκρατικό αλλά το κάνω παρόλα αυτά. Ε, και λέω ότι υπάρχει αυτή η δίκη στην Ισπανία που σημαίνει ότι εμείς πρέπει να περιμένουμε την ετοιμιγορία του δικαστηρίου. Η Μαϊτέ ήθελε το λόγο. Ναι, πολύ πολύ σύντομα. Και εμάς μας ανησυχεί πάρα πολύ το γεγονός ότι αυτή η προστασία μέσω εκκυκλίου είναι πολύ αδύναμη προστασία. Υπάρχει αυτή η νομική διαμάχη. Δεν μας καθυσχάζει αυτό γιατί ε, έχουμε να νομοθετήσουμε για πάρα πολύ λεπτά ζητήματα και ουσιαστικά για πρώτη φορά νομοθετούμε. Και πραγματικά επειδή υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ε, με αυτά που γίνεται. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτά που μας λέτε είναι ικανοποιητικά. Πρέπει από πολιτικές πλευράς να επιβληθείτε περισσότερο ώστε να συγκρατηθεί ε, από τις επαγγελματικές το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν με λάθος τρόπο ε, στοιχεία που έχουν να κάνουν με τόσο σοβαρά θεμελιώδη δικαιώματα. Μάλιστα, λέει ο πρόεδρος. Αυτό ήταν. Τα Δεν μπορούμε ποτέ να καταλήξουμε, κύριε Ιντβελτ. Για να κλείσει η Σοφή. Ναι, έχουμε εκλογέ. Και πρέπει να εξηγήσουμε στου ψηφοφόρου γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλή. Τι καλό κάνει τέλο πάντων. Ήμουν όθηση συγκεκριτήρια για τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων. Πάρα πολλέ ώρε παταλήσαμε για το νομοθέτημα αυτό. Και τώρα τι βλέπουμε, ότι ίσως ε, το καταχρώνται κάποιοι ε, για, τα πολιτικά κόμματα, να αποκομίσουν κάποιο Δεν νομοθετήσαμε για αυτό το λόγο και καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείτε από μόνο σας να το αλλάξετε. Οι επίτροποι θα πρέπει να λάβουν την ευθύνη, αλλά αν το μόνο που μπορεί η Κομισιόν να κάνει όταν υπάρχει κίνδυνο σε παραβίαση Δημοκρατία είναι να σηκώνει τους ώμους και να λέει Του είπαμε ε, ότι δεν μας αρέσει αυτό που κάνετε και αρκεί αυτό είναι ανησυχητικό. Κοντεύει και το τέλος της θητείας. Μάλλον κανείς δεν έχει όρεξη να κάνει και πολλά. Αλλά τόσο δεν προσέχουμε με τη δημοκρατία. Το κάναμε τεχνοκρατικό το ζήτημα. Είμαστε μόλις πέντε βουλευτές εδώ. Είναι πολύ ανησυχητικό. Α, έξι είμαστε. Ω, συγγνώμη. Ναι, κοιτάξτε, πρέπει να φύγω, ε, βιάζομαι. mentioning something. tomorrow or today? carry on. Yeah, carry on. Ναι, συνέχισε. Μήπως να γράψετε στην Κομισιόν Πρόεδρε και να πείτε ότι δεν είμαστε και τόσο ικανοποιημένοι με την αδρανιά τους. Ωραία, θα το ακούσω αυτό. Μιλάμε για το Βασίλη της Ισπανίας τώρα. Είναι και ένα πρόβλημα για μένα. Το Βασίλη της Ισπανίας μου δημιουργεί προβλήματα. 11 Απριλίου έχουμε την τελευταία μας συνεδρία Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει γιατί εγώ έχω να φύγω. Κάποια στιγμή πρέπει να φύγω. Αύριο θα το συζητήσουμε το δικό σας το θέμα. Ωραία. Άρα, 11 Απριλίου είναι η επόμενη και τελευταία συνεδρία της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ στο πλαίσιο αυτής της θητείας. Μήπως και ε, σας απασχολεί αυτό. Αυτή είναι η τελευταία μας συνεδρία, 11 Απριλίου. Καλό βράδυ.